Με μεγάλη μας λύπη ακούσαμε ότι ο Τζανλούκα Μπονάνο ε, ξαφνικά απεβίωσε ο συνάδελφος Μπονάνο έγινε ε, στην θητεία του 2014 μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας καθώς και μέλος της αντιπροσωπείας με τις χώρες ΑΚΕ. Ο κύριος Μπονάνο χθες έπεσε θύμα ενός ε, τραγικού τροχαίου και απεβίωσε στη στιγμή. Ήταν επί σειρά ετών ε, δήμαρχος της Ποροζίζιας στην Ιταλική κοινότητα, του Ιταλικού Δήμου. Η σύζυγός του επεβίωσε, επιβίωσε και ο κ. Μονάνα αφήνει πίσω του γυναίκα και παιδιά. Αυτή η τραγωδία τάραξε βαθιά πολλούς από εμάς και αυτές τις δύσκολες ε, ώρες θέλουμε να εκφράσουμε την ε, συμπαράστασή μας ε, στην γυναίκα του, στην οποία ευχόμαστε και περαστικά και στην οικογένειά του. Σας παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού